Uh, Γεια σας, καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης. Είμαστε λιγοστοί. Ελπίζουμε κι άλλα μέλη να έρθουν πριν την ψηφοφορία. Έχουμε προβλήματα στο Κοινοβούλιο. Ξέρετε με τα συστήματα πληροφορικής. Uh, Και Εν μέρη αυτό είναι ο λόγο που είμαστε ελάχιστοι παρόντε. Ε, Έχουμε προβλήματα να, να αποστείλουμε πληροφορίες στα μέλη, η επικοινωνία είναι δύσκολη. Ελπίζουμε να επιληθεί το πρόβλημα. Ξεκινάμε και ελπίζουμε να έρθουν περισσότερα μέλη όταν θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες με την εξαίρεση φιλανδικών, Λετωνικών, λιθουανικών, μαλτέζικων, βουλγαρικών και κροατικών. Και μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, έτσι. Ωραία, εγκρίνεται. Ανακοινώθηκαν οι γλώσσες τις οποίες έχουμε διερμηνία. Πάμε στο σημείο 3 της ημερησίας διατάξεως για τις υπηρεσίες, για τις δεξιότητες και τα προσόντα, τα επαγγελματικά. Μόλις τώρα ξεκίνησαν οι συζητήσεις και το βασικό θέμα για το Europass είναι ότι παρουσίασε μια νέα δομή το Συμβούλιο για το Europass. Θέλουμε να το αναλύσουμε το θέμα σε τεχνικό επίπεδο, να δούμε ποιες διαφορές υπάρχουν όσον αφορά το περιεχόμενο μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πληροφορίες και γίνονται συζητήσεις με το προσωπικό να πληροφορηθούμε για να συζητήσουμε επί του πολιτικού περιεχομένου του Europass του ε, τούτου λεχθέντος θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαν είναι εισηγητής μπορείτε να μας διαφωτίσετε σας παρακαλώ ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε λοιπόν έχουμε συντάξει μια έκθεση για την Επιτροπή απασχόληση. Συνεργαστήκαμε με την Επιτροπή απολιτισμού, κοινό εγχείρημα. Οικοδομήσαμε καλές γέφυρες με την άλλη Επιτροπή, με τον κύριο Μαλίνοφ. 21 Ιουνίου διεξήχθη ψηφοφορία και ήταν αρκετά πιστικό το αποτέλεσμα 69 υπέρ. Τέσσερις αποχές, μία ψήφος εναντίον. Άρα πήραμε τη διαπραγματευτική εντολή. 64 υπέρ τη εντολής, 6 εναντίον και 2 αποχές. Έλαβε χώρα πρώτος τριμερής διάλογος υπό την ηγεσία της Μαρίτα Όσκοκ, της Προέδρου, που έκανε μια έξοχη δουλειά. Ε, είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε ότι χρειαζόμαστε σύγχρονα εργαλεία που θα εξασφαλίσουν την επίτευξη αποτελεσμάτων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των προσώτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι ομάδες χρησιμοποιούν ε, το Europass, οι εργοδότες, αυτοί που μελετούν, οι επιχειρηματίες οι οποίοι λένε σημειώνουμε αυτά που κάνει η Ευρώπη και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά που μας προσφέρει η Ευρώπη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης ότι αυτές οι δεξιότητες και τα προσόντα ε, θα έχουν τυποποιηθεί και θα γίνουν σεβαστά παρομοίως παρού, παντού συγγνώμη, ε, υπάρχει τμήμα ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει διαφορετική θέση από εμά. Διαφέρει η θέση μα από αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το Europass θα εξακολουθεί να λειτουργεί επί εθελουσία βάσεω. Έτσι πρέπει να παραμείνει. Το ίδιο ισχύει και για το EQF. Ήμουν εισηγητή του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το EQF είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο των Δεξιοτήτων και Προσόντων. Έτσι θα σεβαστούμε τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών, αλλά χρειαζόμαστε και ένα εργαλείο που θα βοηθήσει ε, τη διαφάνεια. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έλαβε χώρα στις 10 Οκτωβρίου. Οι θέσεις ήταν σαφέστατες. Υπήρχε κοινή γραμμή μεταξύ της δικής μας Επιτροπής και της Επιτροπής Πολιτισμού. Τονίσαμε τα βασικά μας θέματα Θέλουμε καταρχάς ε, μια, έναν εξυγχρονισμό της εργαλειοθήκης μας. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τα προσόντα, τις δεξιότητες και τις γνώσεις γενικά. Και ήρθε πια ο καιρός να γίνουν και άλλα βήματα πρόοδου. Τα τελευταία μέτρα υιοθετήθηκαν το 2004. Οπότε τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν θέλουμε όμως ένα εργαλείο, ένα μέσο το οποίο θα είναι πολύ ριζοσπαστικό, θέλουμε εξέλιξη επί των υπαρχόντων. Ο κ. Μάλινοφ δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, αλλά ξεκαθάρισε ότι είναι σημαντικό οι δεξιότητες και τα προσόντα να είναι κάτι που θα δημοσιοποιούν ε, τα κράτη-μέλη, να γνωρίζει ο κόσμος για αυτά. Οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις να τα δέχονται αυτά τα στοιχεία. Διότι όταν αρχίσει η αποδοχή αυτών θα έχουμε πραγματικά ένα χρήσιμο εργαλείο. Η Μαρίτα Ε, το εκπροσώπησε και την αστυνομική κυβέρνηση και τις θέσεις της κυβερνήσεως αυτής στον τριμερή διάλογο και πετύχαμε τέλος Σεπτεμβρίου μια γενική συμφωνία στο Συμβούλιο. Εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι οι διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν είναι πολύ μεγάλες. Συζητήσαμε κάποια άρθρα από το 1 και 2 που εξέτασε ο κ. Μάλινοφ, δηλαδή την ανάγκη να όλα αυτά να εφαρμόζονται επί θελοντικής βάσης. Είναι σημαντικότατο το άρθρο 3 πρόκειται περί των συστημάτων πληροφορικής και ενημέρωσης άρθρα 4 και 9 προστασία των δεδομένων πρέπει να εγγυηθούμε ότι παρέχεται προστασία στα δεδομένα εγώ σχολήθηκα με το άρθρο 5 για τα προσόντα του Europass αυτό σημαίνει ότι οι αρχές πιστοποίησης στα κράτη-μέλη οι επαγγελματικοί φορεί θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν. Όσον αφορά την ΕΣΚΑ, και αυτό είναι σημαντικό για μας, είναι κάτι που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς σαν Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά δεν είναι βάση για περαιτέρω εργασίες. Είναι που, κάτι που δεν είναι γνωστό αυτό στα κράτη-μέλη σαν μέσο. η κεντρική προσέγγιση δεν είναι σωστή. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στη διαδικασία. Τα άθρα 7 και 8 αφορούν την εφαρμογή και τον έλεγχο των μέτρων, υλοποίηση και έλεγχο. Θέλουμε το Europass να είναι διαθέσιμος, διαθέσιμο σε όλους, σε ανθρώπους με αναπηρία, Φερρυπίν. Άρα χρειάζεται μια πολύ ισορροπημένη και συνετική προσέγγιση. Το Συμβούλιο θέλει νέα δομή, εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά αυτό, Για το Άρθρο 6 το ΕΣΚΑ, αυτό καλύπτεται. Άρθρο 11, σύμπραξη με τα κράτη-μέλη, όσον αφορά τις δομές άρθρο 14 και αυτό εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Αφορά και αυτό την υλοποίηση των μέτρων. Σε 9 Νοεμβρίου θα γίνει ο δεύτερος τριμερής διάλογος και νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά προετοιμασμένοι για αυτό το διάλογο. Υπάρχει ευρεία συμφωνία επί πολλών σημείων μεταξύ κρατών μελών, αυτό είναι καλό και θα χρειαστούν και άλλες επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα γίνουν τεχνικής φύσους ε, συναντήσεις 24 Οκτωβρίου, η δεύτερη συνεδρίαση των Σκιωδών, 7 ε, στις 9 Νοεμβρίου μάλλον θα γίνει ο τριμερής διάλογος και 7 Δεκεμβρίου ο τρίτος τριμερής διάλογος. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλή συμφωνία διότι επί των βασικών αρχών δεν έχουμε μεγάλες διαφορές και όσον αφορά τις νέες δόμες, θα επανέλθω και θα σας ενημερώσω την επόμενη φορά. Είναι καλή ατμόσφαιρα, θα το επιβεβαιώσει αυτό και η Πρόεδρος. Είπαμε ότι μπορούμε να δεχθούμε τις διάφορες δομές, δεν έχουμε πραγματικά προβλήματα όσον αφορά τις του Συμβουλίου. Κινούνται σωστά και τα κρατη Είναι καλή η βάση αυτή που υφίσταται και πιστεύω ότι η Ευρώπη θα εγκρίνει κάτι το οποίο τελικά θα είναι ένα μέσο επιτυχές. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Πράγματι επιβεβαιώνω αυτό που είπατε. Πραγματικά ήταν μια πολύ καλή αρχή των συζητήσεων αυτή με τους διάφορους φορείς του συστήματος. Υπάρχει και κάποιος άλλος που έχει συμμετάσχει στις εργασίες που θέλει να πει κάτι. Δεν υπάρχουν και πολλά μέλη παρόντα. Ίσως να παρακαλέσω την κυρία Γιούλτσακ, που είναι υποδιευθύντια μονάδα τη Γενική Διευθύνσεω Απασχόληση, υποτμήματάρχη μάλλον, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Απηχώ το μήνυμα αυτό που ακούστηκε την κακή συνεργασία και σε τεχνικό επίπεδο. Σημειώνεται πρόοδο. Και ευχαριστώ τον συνάδελφο Βίλιαμ που είναι πηγή γνώσεων όσον αφορά το Europass. Με τα χαρά να δώσουμε όση, όση βοήθεια θέλει η γραμματεία του Κοινοβουλίου να παράσχουμε τι αναγκαίε πληροφορίε και σχόλια πως άλλαξε το κείμενο την αρχική πρόταση σε αυτή που έχουμε τώρα επιτάπητος βάσει του σχεδίου κειμένου του Συμβουλίου και επίσης, πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να κινηθούμε σωστά οι συνομοθέτες σε όλο αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Οπότε πάμε στο σημείο 4 της ημερησίας διατάξεως. Ξεκινάμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Υποθέτω ότι δεν θα έρθουν και άλλα μέλη, δεν θα καταφτάσουν και άλλα μέλη. Όπως προανέφερα έχουμε προβλήματα στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε προβλήματα τεχνικής φύσεως και έτσι δεν μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή μέσω μηνυμάτων με τα μέλη. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία. Σε 7 λεπτά θα ξεκινήσουμε. Θα περιμένουμε μέχρι να πάει 9.30. Διότι αυτό προβλεπόταν γραπτός. Χαλαρώστε για 7 λεπτά και θα τα πούμε στις 9.30. Καθίστε παρακαλώ να ξεκινήσουμε φίλοι μου την ψηφοφορία. Πρώτη ψηφοφορία αφορά τη γνωμοδότηση για την κινητοποίηση ε, του Ταμείου για, το, για την Αλμαβίβα, Ιταλία. Θα ψηφίσουμε όλες τις παραγράφους του σχεδίου επιστολής εκτός από την παράγραφο 4 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι για το Ταμείο Προσαρμογής της Παγκοσμιοποίησης, των Πατασμών της Παγκοσμιοποίησης. Ψηφίζουμε την παράγραφο 4 του ΕΛΚ υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός που ξεκινάει τώρα πέρας εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ Το βλέπετε στις οθόνες σας. Υπέρ με 22 ψήφους. Υπέρ. Άρα εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται με 33 ψήφους. Πάμε στη συμβαστική 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για αυτούς που ήρθαν αργά, καθυστερημένοι, για την εφ εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενώσης για ε, την αναπηρία, τροπολογία συμβαστική 2, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 101, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 102, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 102 άρχεται η ψηφοφορία πέρας αυτής εγκρίνεται με 15 ψήφους τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασ... ε, η τροπολογία συμβιβαστική 5 υπέρ Καταπίπτει, διότι τροπολογία 119 νεκρήθη. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 123 με την 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Amendment 145 υπέρ. Όχι, δεν έχει. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Those against, abstentions... Κατά αποχές εγκρίνεται. το πολύ 153 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 158 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 172 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Amendment Τρομολογία 176 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 177 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 179 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 180 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 185 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 186 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά έλεγχος για τη συμβαστική 12 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται με 24 ψήφους συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για την τροπολογία 209 ξεκινάμε τώρα πέρας και εγκρίνεται με 17 ψήφους συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά έλεγχος για τη συμβαστική 20 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους. Προχωρούμε. Τροπολογία 232. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 233. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 234 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά δεν βλέπω τι γίνεται με την 21 τη συμβαστική ξανά 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 244 υπέρ όχι λέει πρόεδρος ναι 244 μαζί με τη 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 249 όχι, δεν την ψηφίζουμε. Τροπολογία 251 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 252 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για τη 252. Ξεκινάμε τώρα την ψηφοφορία. Πέρας για τη 252 εγκρίνεται με 28 ψήφους. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 275 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 277 υπέρ κατά άποχες Ας ελέγξουμε τη 277. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 27 ψήφους. Τροπολογία 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κολτ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κολτ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κολτ 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κολτ 12 υπέρ κατά το πρώτο τμήμα Απ' την αρχή, πάμε ξανά. Κολτ 12, πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε λοιπόν την Culture 12, πρώτο τμήμα της Επιτροπής Πολιτισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους. Πάμε στην κολ 17 λέει η Πρόεδρος. κολ COP17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρινεται κόλ COP23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κολ 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 288 Συγγνώμη, λέει 289 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 290 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για τη 290 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται με 25 ψήφους συμβιβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 295 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την NV34, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 24 ε, ψήφους. NV36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV340 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 37 Συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 317 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 318 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «321», τροπολογία 321, θα ψηφιστεί, όχι με συγχωρείτε λέει η πρόεδρος, είναι εκτός πεδίου. Άρα συμβαστική 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 323 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 324 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 325 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 331 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 332 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 339 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 πετή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 341 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 346 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 350 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται λέει η πρόεδρος. Ας επαληθεύσουμε. 350 αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Και εγκρίνεται με 27 ψήφους. 351 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 352 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 353 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 354 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 355 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 357 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 365 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 366 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 377 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 387 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 400 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 405 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 406 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πετή 30 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Επαλήθευση, καλώς πέτει, δηλαδή επιτροπή Αναφορών, υπαριθμούν 30. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Απερίφθη με 24 ψήφους. Συμβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 419 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 420 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 421 μαζί με την 399 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 422 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 424 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 425 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 426 εκπίπτει. Πετή 1. Πρώτο μέρος, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΠΕΤΗ 2, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Ας επαναλάβουμε. Πέτη 2, δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Πέτη 5, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Πέτη 6, υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Πέτη 18, υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Πέτη 38, υπέρ κατά. Ε,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 Συμβαστική 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 και 33 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 36 και 37 ομοίως υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40, συγγνώμη, συμβιβαστική 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 αυτή όμως καταπίπτει. Άρα ακολουθεί 74 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ είναι ίδια. Καλώ. Τότε τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 σημαντική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 και 72 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 86 μαζί με την 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 εκπίπτει 89 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. NVV υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. NVD δέλτα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. NV, α, δεν ψηφίζουμε την Age. πηγαίνουμε στην NVI, δηλαδή γιώτα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε Αρχίζει η ψηφοφορία που είναι ονομαστική. Αρχίζει λοιπόν. Τέλος τώρα. Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ και καμία κατά. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Now we are on the next... Η πρόεδρος. Προχωρούμε στην επόμενη ε, λίστα ψηφοφορίας, διότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη και απασχόληση. Αρχίζουμε με τη συμβαστική Α. Σημειώνω ότι η συγητής είναι ο κύριος Λόπεθ. Συμβαστική Α, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Της τροπολογίας 140 θα ψηφιστεί ως προσθήκη στην συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is now. Τέλος της ψηφοφορίας. And it's carried by Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ. Η ε, συμβαστική ΚΑΠΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΔΕΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 157 υπέρ κατά αποχές λέω πως απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 157. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 159. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλλά νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Οπότε άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. Απορρίπτεται με 23 ψήφους. Πάμε στην συμβιβαστική L. Ονομαστική κλίση ε, έχει ζητήσει, έχουν ζητήσει οι 11 persons must be in favor of this. 11 πρέπει να είναι υπέρ. Ωραία, είστε 11. Ωραία, θα κάνουμε λοιπόν ονομαστική για την ε, συμβιβαστική L. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is now closed. Τέλος. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. Compromise M, those in favor. Ε, υπέρ, κατά, αποχές για τη συμβαστική M. Ε, ε τώρα η νη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Compromise P, Συμβιβαστική P. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R, ρο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Compromise Συμβεβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 205 κατά τμήματα ψηφοφορία το έχει ζητήσει το ΕΛΚ. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική W. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. α, ΑΑ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3β. Ονομαστική έχει ζητήσει, έχουν ζητήσει οι σοσιαλιστές. They are still 11. Uh, ε, yes. So, uh, yes. So we vote, uh, we take a roll call vote on Ονομαστική λοιπόν ψηφοφορία για την πρώτη συμβαστική 3 β, ΒΒΒ. β, β. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο Τώρα κάνουμε ονομαστική πάλι κλίση για τη συμβαστική β, β. Εντάξει και πάλι στα 11, ωραία. Ονομαστική άρχεται για την ΒΒ. Τέλος. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες και αρχίζουμε με την 224, 225 και 226 που είναι ταυτόσημες. Υπέρ, κατά, αποχές, Κρίνονται νομίζω. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται και κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην συμβιβαστική CC. Υπέρα κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική DD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, τροπολογία 243 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε τη 243 δεν βλέπω άρχεται η ψηφοφορία και τέλος τώρα της ψηφοφορίας για τη 243. Απορρίπτεται με 24, 24 ψήφους. Μετά έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία από το ΕΛΚ για τη 244, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική ΕΕ. Ονομαστική ψηφοφορία έχουν ζητήσει οι σοσιαλιστέ. Εντάξει, ακόμα 11 είστε. Κάνουμε λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία για την ΕΕ. Άρχεται. Τέλος τώρα της ψηφοφορίας. And it's carried by three votes. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους διαφορά. Okay. We go to compromise FF on... Πάμε στη συμβιβαστική φουφού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική GG. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Compromise HH. Uh, roll call vote. Συμβιβαστική HH. Υπέρ κατά αποχές. Αυτό, εδώ αρχίζουμε και ψηφίζουμε ε, ονομαστική ψηφοφορία για την HH. And, uh, the vote is now clear. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ. Προχωράμε στην 3H. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 271. Η πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 271 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 274 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε για τη 274 και άρχεται η ψηφοφορία, τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 26 ψήφους. 275 Ποιοι είναι υπέρ της διαγραφής της 275 Κατά Πρέπει να ελέγξουμε εδώ Οπότε ελέγχουμε. Πρόκειται για τη 275 που θέλει να διαγράψει. Τέλος. Μάλιστα. Πάμε σε, εγκρίνεται και πάμε κατευθείαν στην συμβιβαστική 2. Α, όχι, συγγνώμη. Ποιοι είναι υπέρ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική J, J. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική K, K. κάπα κάπα Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 293. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 294 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική LL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική MM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική νι νι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον όμικρον. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 326. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα κάνουμε κατά τμήματα ψηφοφορίες για την 327. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, αλλά ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται, τέλος, απορρίπτεται με 26 ψήφους. Συμβιβαστική πι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική QQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 345 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ρορό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική SS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 2, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τι; Τι; ε, ταφ ονομαστική, ζήτησαν οι σοσιαλιστές. Είστε ακόμη 11 εδώ, μάλιστα, ωραία. Αυτό σημαίνει ότι ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται για την ε, συμβαστική ΤΑΦ. ΤΑΦ τέλος της ψηφοφορίας και εκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ. Συμβιβαστική 6-6, χ, χ, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραπολογία 361, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική U, Προτείνεται ονομαστική κλίση από τους σοσιαλιστές, οπότε ψηφίζουμε, άρχεται. And the vote on compromise UU is now closed. Τέλος. Απορρίπτεται με 27 ψήφους. Προχωράμε λόγω αυτού στην τροπολογία 363. Υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 363 ε, άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται We'll go to amendment 370. Those in favor, those 370 υπέρ κατά αποχές λέω πως απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε and the vote is open and... τέλος ψηφοφορίας και... απορρίπτεται we go to amendment 369 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 369 άρχεται πέρας εγκρίνεται με 23 ψήφους πάμε στην τροπολογία 373 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική VV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το αρχικό κείμενο παράγραφος 31 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την παράγραφο 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 23 ψήφους. Τροπολογία 380. Το, το ΕΛΚ ζήτησε κατά τμήματα ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά Εγώ θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική WW υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική YY υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 389 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεν ψηφίζουμε την 390 πάμε συμβαστική ζήτα ζήτα υπέρ κατά έλεγχος όσον αφορά την ζήτα δεν είναι σαφής η αντιδράσεις άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβατική ZZ η ζήτα ζήτα πέρας απορρίπτεται με 23 ε, ψήφους. We go to amendment 391, those in 391 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για την 391 άρχεται η ψηφοφορία πέρας για την 391 εγκρίνεται με 25 ψήφους τροπολογία 394 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 394 έλεγχος άρχεται πέρας εγκρίνεται με 22 ψήφους. Τροπολογία 395 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 395 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με 25 ψήφους. Συμβαστική ζήτα α υπέρ κατά Συγγνώμη, πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την Ζ ZA. Πέρας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους. Συμβαστική ΖΒ υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται έλεγχος για τη συμβατική, συμβαστική συγγνώμη ΖΒ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους. Τροπολογία 400 υπέρ. Αποχές. Uh, uh, Έλεγχος για 400. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 24 ψήφους. Τροπολογία 401 και 402 καταπίπτουν. Συμβαστική ZC υπέρ κατά αποχές. Ε, που 10 υπέρ κατά αποχές. Εγώ λέω ότι μάλλον εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την τροπολογία 10. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρινέται με 22 ψήφους. Πάμε στην τροπολογία 16 στις ιδεολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το συμβαστική Αλφαβήτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οίκον C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται συγγνώμη. Συμβαστική ΕΗ e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές α, έλεγχος για την 38 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με 24 ψήφους τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική αι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ΑΚ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική αλφα μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τοπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για την τροπολογία 54 άρχεται η ψηφοφορία για την 54 πέρας εγκρίνεται με 22 ψήφους τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την τροπολογία 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 22 ψήφους. Τροπολογία 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 67 υπέρ κατά έλεγχος για την 67 άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με 21 ψήφους 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική α όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έλεγχος για την 79. Ξεκινάει τώρα η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 22 ψήφους. Τροπολογία 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο της τροποποιημένης έκθεσης με ονομαστική ψηφοφορία που άρχεται τώρα. And the vote is now closed. Πέρας. 37... 37 ψήφοι υπέρ. Και ευχαριστώ τον εισηγητή για το δουλειά που έκανα. Okay. We will soon proceed with Mr. Θα προχωρήσουμε σε λίγο με την έκθεση του κύριου Λαβελέ. Ένα λεπτό για να αποχωρήσουν όσοι θέλουν με ησυχία από την αίθουσα. We proceed. We proceed.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 χρηματοδοτιστικοί κανόνες που αφορούν το γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ε, ε, ε, Ψιθυριστά αν μπορείτε να συζητήσετε. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Mr. Lavrille, are you... Κύριε Λαβελέ, Είστε έτοιμος να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Έχετε το λόγο. Ησυχία στο ακροατήριο παρακαλώ. Ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι σύντομο. Μετά τη ψηφοφορία στην Επιτροπή του Σχεδίου Γνωμοδότηση για του του κανόνε που ισχύουν για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, Omnibus, δηλαδή το συνολικό αυτό έργο που η Επιτροπή επασχόληση η αποκλειστική αρμοδιότητα, το FSF, τα τέσσερα ταμεία και το πρόγραμμα EASY ε, ξεκίνησα τις διαπραγματεύσει για τις οποίες μου δόθηκε εντολή ε, στον τριμερή διάλογο και σήμερα σας λέω πώς πήγαν οι διαπραγματεύσει. Ε, ε, πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις ε, τριμερής ήταν καρποφόροι, καταλήξαμε σε συνένεση στα πλαίσια της εντολή που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τελικά συγκεράστηκαν κάποιε απόψει Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δικέ μα. Είμαστε στα μέσα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Θέλαμε να προστεύσουμε του εφαρμοστέ κανόνε και να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα ταμεία. Πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσει ε, πηγαίνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Ήδη έχουμε συμφωνήσει επί κάποιων σημείων στον τριμερή διάλογο. Βέβαια απομένουν κάποια σημεία σημαντικά προ ρύθμιση, αλλά έχω την πεποίθηση ότι ο επόμενο τριμερή διάλογο, ο οποίος θα λάβει χώρα κανονικά αρχέ Νοεμβρίου, θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις. Ε, μπορώ να σα πω περισσότερα αν θέλετε. Ε, θα μπω σε λεπτομέρειε αν το θέλετε, ακόμα και αν το θέλετε. Ε, όσον αφορά το FSC, συμφωνήσαμε τα τρία μέρη. Όσον αφορά τον ορισμό, τα κριτήρια που θα είναι κειμενικά όσον αφορά τι επιδόσεις των προγραμμάτων, επάνω Έχουμε ξανά την κατανομή του προπολογισμού που θα είναι αντικειμενικά κριτήρια που θα ακολουθούνται κατόπιν αιτήματο των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων. Επίση, έχουμε καταλήξει συμφωνία, αν συμπεριλαμβάνουμε στον κανονισμό, μία αναφορά στου κοινού κανόνε για όλα τα ταμεία. Ούτω ώστε οι δύο κανονισμοί ε, να έχουν ε, συγκεκριμένε αναφορέ δικαιούχου. Αυτό είναι θετικό, πιστεύω. Όσον αφορά τα εκρεμή σημεία στι διαπραγματεύσει, περιμένουμε ακόμα κάποια προτότηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωση όσον αφορά τι ενδεχόμενε παρεκκλήσει από τον κανόνα των ελάχιστων προδιαγραφών de minimis. Μετά την πρόταση που έκανα και που επικυρώσατε εσεί, να ανέβει στα 150.000 ε, ευρώ το ανώτατο όριο ετέφεση ε, έχουμε καταλήξει, πλησιάζουμε σε συνένεση που ολοκληρωθεί στον τελικό του διάλογο και θα πρέπει η δημόσια υποστήριξη να πάει στα 150.000 ευρώ μόνο για το FSE και την περίοδο την διετή που αφορά το κείμενό μας και 100.000 για τα άλλα ταμεία. Όσον αφορά το FAD, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα διατύπωσης που δεν είναι παντού η ίδια στον κανονισμό και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ερμηνείας. Αλλού χρησιμοποιείται αναστολή και αλλού διακοπή. Ο Ρώσο όσον αφορά τι πληρωμέ που καταβάλλονται στα κρατη Η συμφωνία που τελικά πετέφθη μεταξύ των τριών μερών ήταν να θυμηθεί η διατύπωση επί αναστολή, εισάγοντα τον ορισμό του όρου στον κανονισμό για περισσότερη σαφήνεια. Όσον αφορά το FME, συμφωνήσαμε για μια διατύπωση σωστή όσον αφορά την εφαρμογή του FME σε ομάδε ομίλου επιχειρήσεων και θέλουμε να ισχύει για επιχειρήσει που συμμερίζονται τον ίδιο τομέα, μοιράζονται την ίδια περιφέρεια. Νομίζω ότι είναι μια πρόοδο εξαιρετικά σημαντική που θα επιτρέψει να μην ε, είναι αυτό το ταμείο μόνο για του μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων. Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των περιφερειών με ένα επίπεδο ανεργία ε, νέων υψηλό, η διατύπωση που συμφωνήσαμε στην τριμερή διάλογο θα πρέπει να καθορίζει να είναι 20% το επίπεδο τη ανεργία σε σχετικά με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και αυτή είναι μια άποψη ε, που ε, ερμηνεύεται ανάλογα με τη χώρα. Μετά όσον αφορά το πρόγραμμα EASY, το πρόγραμμα EASY και το πώς κατανέμεται ο προπολογισμό όσον αφορά τους τρεις άξονες, ΕΡΕΣ και μικροχρηματοδότηση και διάφορους τομείς θεματικούς που ανήκουν στο σημείο που διαπραγματευόμεθα ακόμα μέχρι τώρα. Ε, ελπίζω και πιστεύω εξάλλου ότι είμαστε κοντά σε μια συνένεση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε αρκετά γρήγορα στη συμφωνία από αυτού. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο πρότεινε ένα ποσοστό τουλάχιστον 45% για το Progress και το 18% για τους δύο άλλους άξονες. Αυτή είναι μια πρόταση που προσεγγίζει τις δικές μας, αλλά ακόμα και αν προσεγγίζει όμως ε, απέχουμε αρκετά. Πιστεύουμε ότι είναι ένα ποσοστό πολύ χαμηλό ακόμα, αλλά λαμβάνοντα υπόψη την εντολή που μας έχει δοθεί. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσει και θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε τα επιχειρήματα τους ώστε να πείσουμε τους συνομιλητές μας. Ιδού λοιπόν ποια είναι η κατάσταση των διαπραγματεύσει που συνεχίζονται στον φατική νομοδότηση να διευκρινίσω ότι όπως μπορείτε να δείτε σεβαστήκαμε την εντολή που μας ανετέθη από την Επιτροπή Απασχόλησης. Λοιπόν, η συμφωνία τελική του μερίου διαλόγου στην Επιτροπή Απασχόληση θα ψηφιστεί πριν υποβληθεί στην Ολομέλεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλου ιδιαίτερω του σκιώδεις εισηγητέ, εκείνους τουλάχιστον που συνάντησα, οι οποίοι βοήθησαν και με βοηθούν ακόμα για την σωστή ομαλή εξέλιξη των πραγματεύσεων, Πυρίνσκι και Σελίμοβιτς ιδίω. Τους ευχαριστώ θερμότατα. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συνεργάτες των ομάδων και τους συνεργάτες μου που κάνουν φανταστική δουλειά βοηθώντας με όσον αφορά την πρώτη μου έκθεση και τον πρώτο μου τριμερή διάλογο στην ε, καριέρα μου αυτή τη νέα που έχω ε, στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω όλες τις απαντήσεις. Αν δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σήμερα θα σας τις στείλω στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Λαβελέ. Πάντοτε υπάρχει μια πρώτη φορά. έχουμε να ασχοληθούμε με τόσο διαφορετικά θέματα που πάντα είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. I'll give the floor to uh, uh, Mr. Madam Chair, I have nothing uh, in particular to add. I would also... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να πω πολλά. Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για τον τρόπο με τον οποίο ε, έκανε την εργασία ο εισηγητής και τη συνεργασία που είχαμε μαζί. Ευχαριστώ. Is Madame Trebesius here? No. Trebesius είναι εδώ. Όχι. Mm. Σελίμοβιτς. Ούτε. Πιμέντα Λόπες επίσης. Βάνα. Η Μόνικα Βάνα όχι. Και εσείς δεν αντικαθιστάτε κανέναν. Και ούτε και ο κύριος Ντομινίκ Μαρτά. Έχουμε κάποιον από την Κομισιόν. Yes, Madam Fellay, Please. Ναι, η κυρία Fellay. Thank you, Mrs. Chairman. Uh, on the Commission side, we would just like as well to thank the rapporteur and the whole uh, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλη την ομάδα του Κοινοβουλίου ε, για την καρποφόρα συνεργασία. Είμαστε βέβαιοι ότι με μικρή προσπάθεια θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις την επόμενο τριμέρι και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε σε συμβαστικές. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Λαβελέ. Εξαντλήθηκαν ε, οι συνάδελφοι μετά από τις ψηφοφορίες και είμαστε πιο μπροστά στην ημερησία μας διάταξη. και ένα σημαντικό θέμα στην ημερήσια μας διάταξη. Δεν είμαι βέβαια ότι το γνωρίζετε όλοι επειδή το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. για να στείλει τα μηνύματα σε όλους. Αλλά στις 11 και 4 θα έχουμε μια παρουσίαση play on social... της κατάστασης προοδού για το θέμα της διακήρυξης του κοινωνικού πυλώνα Πολλά ζητήματα λοιπόν έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή για αυτό εδώ το ζήτημα. Και είχαμε και μια βαθιά συζήτηση στην τελευταία συνάντηση των συντονιστών μας. Ζητήσαμε από τους δύο Σέρπα, τον κύριο Βαντεκάντελερ και την κυρία Ροντρίγκε να έρθουν στην Επιτροπή μας, αλλά δεν θα είναι εδώ παρά μόνο στι 11 και 4. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα λιγότεροι θα συμμετέχουν στη συζήτηση. Ελπίζω όμως πως κάποιοι από εσάς θα παραμείνετε. Διότι έχει αυτό να κάνει με την εκπροσώπησή μας σε αυτήν τη συνεδρίαση. Βέβαια, εμείς ελπίζουμε ότι η διακήρυξη του κοινωνικού πυλώνα είναι, θεωρούμε μάλλον ότι είναι δική μας αρμοδιότητα εδώ σε αυτήν την Επιτροπή, αλλά η Επιτροπή από ό,τι φαίνεται έχει, δεν έχει καμιά επίσημη εκπροσώπηση. Οι δύο Σέρπα που έχουν επιλεγεί από τον κύριο Ταγιάννη είναι αυτοί που ασχολούνται με όλη τη δουλειά που γίνεται. Θα ήταν χρήσιμο και θα ήταν και σοφό Θα δούμε λοιπόν ποιος είναι αρμόδιος γιατί, στην, ποια είναι η αρμόδια επιτροπή και θα έχουμε τις εκθέσεις αντικάντλερ. Ελπίζω πραγματικά στις 11 και 4 θα είστε εδώ. Κάποιοι από εσά τουλάχιστον. Ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε να στείλαμε και μια επιστολή στον Ταγιάννη με τους συντονιστές και με όλους τους, ε, όλες τις ομάδες γιατί θεωρούμε ότι η Επιτροπή που είναι αρμόδια για τα κοινωνικά θέματα, δεν έχει κάποια επίσημη ατζέντα και δεν έχει προσκληθεί όπως έχουν προσκληθεί αυτοί οι ΣΕΡΠΑ. Ε, λοιπόν, διακόπτουμε τη συνεδρίαση τώρα. Θα συνεχίσουμε στις 11 και 4 και ελπίζω πως αν δεν μπορείτε να έρθετε εδώ, στείλετε κάποιον άλλον που να μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό σας. για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε, όπως το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή ότι η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη και αρμόδια για την κοινωνική ατζέντα να εκπροσωπείται με κάποιο τρόπο στη συνεδρίαση στο Γκέτεμπορκ στις 17 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ και διάλειμμα έχουμε μέχρι τις 11 και 4. Ε, thank ε, Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, που επανήλθατε στην αίθουσα και έχουμε πλέον ολοκληρώσει τις ψηφοφορίες και μάλιστα νωρίτερα από ό,τι είχαμε αρχικά σχεδιάσει. Ε, κάναμε ένα διάλειμμα και καλώς ήρθατε και πάλι στην αίθουσα. Θα προχωρήσουμε στο υπαριθμό 8 της ημερήσιας διάταξης παρουσίαση του State of Play για τον κοινωνικό πυλώνα. Θα αρχίσω πρώτα δίνοντας τον λόγο στους Σέρπα. Ο κύριος Βαντεκεντελάρ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα προχωρήσω με την Μαρία Ζωάου Ροντρίγκες. Κύριε Βαν Κέντελα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, όπως είπε και η πρόεδρος, μας στις 7 Σεπτεμβρίου η κυρία Ροντρίγκε, εγώ και ο Τόμας Χέντελ αναλάβαμε Σέρπας και έχουμε μεγάλη τιμή που μιλούμε ενώπιον σας σήμερα σε μια ε, εφάπαξη διαδικασία για την προκήρυξη ε, του κοινωνικού πυλώνα που έχει μια ιδιαίτερη σημασία και χρειάζεται πράγματι και ειδικέ λύσεις όταν πρόκειται για την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου. Η διάσκεψη των Προέδρων θεώρησε ότι ο ορισμός των τριών ΣΕΡΠΑ είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει για τις 17 Νοεμβρίου, όπως ξέρετε όλοι, ε, στο Γκότενμπουργκ, που θα είναι ιδιαίτερα πολιτικού χαρακτήρα όπου οι ηγέτες θα ε, επαναδιακηρύξουν την πίστη τους ε, στην ανάγκη για ένα κοινωνικό, κοινωνικό πυλώνα κλπ. Και βεβαίω υπό την Εστονική Προεδρία, Προεδρία του Συμβουλίου. Όσον αφορά τον δικό μας ρόλο, τον ΣΕΡΠΑ, νομίζω μιλώ και εξ ονόματος της κυρίας ε, Μαρία Ζωά, παίζουμε το ρόλο μας όσο πιο πιστά γίνεται και βεβαίως και όσο και πιο κοντά στο περιεχόμενο της έκθεσης πρωτοβουλίας που έχει ψηφιστεί και φιλοδοξία των τριών ΣΕΡΠΑ είναι να ψηφιστεί ένα κείμενο το οποίο θα είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο κείμενο της έκθεσης πρωτοβουλίας. Διαπραγματεύσεις. Τρεις ανεπίσημες συναντήσεις τριμερούς διαλόγους. Στην πρώτη το Κοινοβούλιο, η Προεδρία του Συμβουλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν να αφήσουν άθικτες τις 20 αρχές της ε, προκήρυξης, της διακήρυξης καλύτερα. Άρα συζητήθηκε το προήμιο του κειμένου. Ειλικρινά το κείμενο ήταν αρχικά πολύ εξισορροπημένο. Παρ' όλα αυτά ήταν σαφές επίσης εξ αρχής ότι μένουν ορισμένα ζητήματα ανοιχτά για συζήτηση στο Συμβούλιο. Θα σας συζητήσω δύο και μετά βεβαίως θα δώσω το λόγο στην, ε, ε, θα παραδώσω το μικρόφωνο στην κυρία Ροντρίγκε. Το πρώτο ήταν λοιπόν η δημοσιονομική επίπτωση του κοινωνικού πυλώνα. Η δημοσιονομική ισορροπία δεν επιτρέπεται να επηρεαστεί από την διακήρυξη. Και τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν σε μια διατύπωση που ευθυγραμμίζεται με τις συνθήκες και ιδίως το άρθρο 154 που διευκρινίζει ότι προφανώς οι χώρες μέλη μπορούν να διαχειρίζονται τα δημόσια οικονομικά και ότι ο κοινωνικός πυλώνας δεν πρέπει να επηρεάσει την δημοσιονομική ισορροπία. Ένα δεύτερο σημείο ανησυχίας για το Συμβούλιο ήταν το πεδίο εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Και εδώ συμφωνήσαμε επί ενός κειμένου, το οποίο συμβαδίζει με τις συνθήκες και πλησιάζει και στο περιεχόμενο της ε, έκθεσης πρωτοβουλίας και που ξεκαθαρίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του πυλώνα αναφέρεται στις χώρες της ζώνης ευρώ, αλλά βεβαίως επηρεάζει και τις άλλες. Για τα επόμενα δύο θέματα της συζητήσεως, νομίζω υπάρχει άλλο ένα ανοιχτό θέμα, ανοιχτό στι διαπραγματεύσεις, αλλά βεβαίω δεν είμαι και ο μοναδικό ομιλητή, γι' αυτό θα αφήσω τη συνάδελφό μου να μιλήσει. Τέλο όμω θέλω να ολοκληρώσω την ε, πολύ σύντομη αυτή ενημέρωση, λέγοντα σα ότι οι ανεπίσημε συνομιλίε με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα ήταν πολύ ανοιχτέ έω τώρα και από το κλίμα των συζητήσεων θεωρώ ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί η συμφωνία στις επόμενες ημέρες με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. I will then give the floor to Madam... Uh, ευχαριστώ. Ας λάβει το λόγο τώρα η κυρία Ροντρίγκης. Έχω να σα πω και εγώ τα εξή στην Επιτροπή Απασχολήσεως. Αφού σας ευχαριστήσω πρώτα για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας απευθύνουμε το λόγο, διότι εσεί τα μέλη τη Επιτροπής Απασχολήσεως θα πρέπει να είστε πλήρως ενήμεροι για τα τεκτερόμενα. Δεύτερο, όπως είπε και ο συναδελφό μου μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχουν λάβει χώρα επαφέ μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων σε ανεπίσημη βάση με στόχο την διευκόλυνση μια ενδεχόμενη συμφωνίας στις συνεχιζόμενες συζητήσεις μέσα στο Συμβούλιο των Υπουργών. Εγώ θεωρώ ότι ο τριμερής αυτός διάλογος, ανεπίσημος βεβαίως, έπαιξε θετικό και επικοδομητικό ρόλο. Και όπως εξήγησε μόλις ο συναδελφός μου, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Πλησιάζουμε στα συμπεράσματα. Για την σύνταξη της διακήρυξης που θα είναι ένα σημαντικό πολιτικό βήμα η κοινωνική Ευρώπη δηλαδή που αντιμετωπίζει τις νέες κοινωνικές προκλήσεις. Έρχεται η στιγμή αυτή. Θα πρέπει να είμαστε υπερήφανες και υπερήφανοι διότι η έκθεση του Κοινοβουλίου μας με στήριξη πέντε πολιτικών ομάδων το περιεχόμενο της εκθέσης αυτής δηλαδή, απηχείται σε σημαντικό βαθμό στις 20 αρχές της διακήρυξης. Αυτές οι 20 αρχές απηχούν τις αξιώσεις που προβάλλουμε στην εκθεσή μας και εμείς εφόσον αυτές εγκριθούν θεωρούμε ότι κλείνει η διαπραγμάτευση. Σε ό,τι αφορά το προήμιο. Και εκεί επιτύχαμε σημαντική σύγκληση αφενός με την εξασφάλιση του ότι ο κοινωνικός πυλώνας θα ισχύει για όλες τις χώρες μέλη και όχι μόνο για τη ζώνη ευρώ. Γνωρίζετε ωστόσο ότι αυτή ήταν ε, η αρχική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλες οι θέσεις που αναπτύξαμε δημοσία μέχρι τώρα. Δεύτερο, έχουμε και διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά την ανάγκη να ευθυγραμμίζονται αυτά με τις ε, ευρωπαϊκές συνθήκες. Δεύτερο, δημοσιονομική ευθύνη και περιθώριο διαχείριση των εθνικών προϋπολογισμών. Επ' αυτών όλων συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο. Και μας μένει μια δυσκολία τώρα, η οποία δυσκολία αναφέρεται στην δυσκολία που πρέπει, στην, συγγνώμη, στην ε, επιλογή που πρέπει να γίνει για την εφαρμογή του πυλώνα. Πιστεύω ότι είχαμε μια καλή λύση που ανεφεί μέσα από τις διαπραγματεύσεις με τα άλλα δύο θεσμικά οργάνα. Τώρα όμως το Συμβούλιο προτείνει να προσθεθεί μια λέξη που για μας πραγματικά δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή. Ως εξής, στην εξή πρόταση ή φράση. Οι αρχές και τα δικαιώματα για να μπορούν να εφαρμόζονται χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα και νομοθεσία που θα εγκριθούν στο κατάλληλο επίπεδο. Αυτή είναι η διατύπωση στην οποία βασίσαμε τις εργασίες μας. Τώρα το Συμβούλιο προτείνει να μπει η λέξη would require ε, δηλαδή θα απαιτούν ή θα απαιτούσαν κατάλληλα μέτρα και νομοθεσία να εγκριθεί στο κατάλληλο επίπεδο. Να σας εξηγήσω γιατί θεωρώ εγώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιτρέπεται να δεχθεί την διατύπωση αυτή. Πρώτα διότι αυτό το good είναι υποθετική, είναι, ε, εκφράζει τον υποθετικό λόγο. Υποθετικός λόγος, ξαναλέγω. Άρα δεν είναι κατάλληλο για να μπει σε μια διακήρυξη. Μια διακήρυξη δεν μπορεί να χρησιμοποιεί υποθετικό λόγο. Θα πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα, όχι σε υποθέσεις. Υπάρχει και ένα δεύτερο επιχείρημα, ότι δηλαδή εμείς θέλουμε να είναι αξιόπιστος ο ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας. Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινή γνώμης που είναι πολύ υψηλέ. Το μήνυμά μου προ το Συμβούλιο Υπουργών είναι σας παρακαλώ επανεξετάστε το. Διότι όταν θα ξανασυναντηθούμε στην ΕΠΣΚΟ θα πρέπει να μπορέσετε να συμφωνήσετε σε κάτι το οποίο θα κρίνει η κοινή γνώμη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κατάλληλη λέξη για το περιεχόμενο μιας διακήρυξης. Αυτό λοιπόν είναι το ακριβές μήνυμα που στέλνω εγώ ή θα στείλω αύριο στην Κορεπέρ και μετά στην Εύσκο. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί λύση μέχρι την αυριανή συνάντηση των μόνιμων αντιπροσώπων, Κορεπέρ δηλαδή, ώστε να ανοίξουν πλέον οι συνθήκες, να, να, να υπάρξουν οι συνθήκες αν θέλετε για μια αξιοπρεπή εκδήλωση που θα γίνει στο Λουξεμβούργο με σημαντική παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αρκούμε σε αυτά τα λόγια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις από τους παριστέμενους. Ο κ. Κάσα από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχα την ευκαιρία ήδη να το συζητήσω αυτό σε επίπεδο συντονιστών είναι σημαντικό επίσης που διεξάγεται αυτή η συζήτηση τώρα μεταξύ των μελών της παρούσης Επιτροπής. Ευχαριστώ τους ΣΕΡΠΑΣ καταρχάς για το έργο τους πάνω σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα, το sui generis αυτό εγχείρημα, πάρα πολύ σημαντικό όπως είπε και ο Τόμ, είναι μοναδική ευκαιρία που δημιουργείται. Όλοι μας εδώ εργαστήκαμε σκληρά, ούτω ώστε να θεσπίσουμε αυτές τις αρχές που θα τύχουν μεγάλης υποστήριξης από τα θεσμικά όργανα, όλα πιστεύω, και πιστεύουμε ότι δεν θα είναι εύκολο οι πάντες να πετύχουν τα πάντα που θεωρούν ότι είναι καλό να επιτευχθούν. Θα πρέπει να υπάρχει δούνε και λαβήν. Είναι απλώς μια πολιτική δήλωση, μη δεσμευτική. Ανησυχώ για κάτι όμως. Ότι παρόλο που δεν θα μας αρέσει η προτινόμενη διατύπωση σε όλα τα σημεία, ας μην δώσουμε την ευκαιρία σε άλλα θεσμικά όργανα να αρχίσουν να προβάλλουν αντιρρήσεις σε άλλα σημεία, σε διατυπώσεις που θέλουμε εμείς να παραμείνουν. Συμβουλή που σας απευθύνω και στους δύο, για να μην μακρηγορώ, να μιλήσω και άλλοι συνάδελφοι, είναι το εξής να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να νικήσουμε 100% σε αυτή τη μάχη, ας διαπραγματευτούμε με τα άλλα θεσμικά όργανα και δεν πιστεύω ότι μία λέξη θα πρέπει να μας οδηγήσει να πούμε ότι δεν θα αποδεχτούμε ποτέ το κείμενο. Ας διαπραγματευτούμε. Ας είμαστε πιο γενναιόδοροι. Ας συμφωνήσουμε με όλα τα θεσμικά όργανα, ούτω ώστε αυτή η μοναδική ευκαιρία να μην χαθεί. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο, όλο ιδιαίτερο στο Συμβούλιο, να τους δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε και θέλουμε να περάσει αυτό. Ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Ξέρω ότι έχετε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά σας τι επόμενες ημέρες. Παρακαλώ προσπαθήστε να είστε πιο γενναιόδοροι όσον αφορά ε, τι που έχει το Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Ευχαριστώ κύριε Κάσα. Η κυρία Γιουγκέριου έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Ξεκινώντα θέλω να ευχαριστήσω του Σέρπας για τη δουλειά που έκαναν μέχρι τώρα. Παρόλο που συνήθως είμαι πολύ γενναιόδορη, αυτό πιστεύω, σε αυτή την περίπτωση έχω κάποια ερωτηματικά που μου δημιουργούνται. Είναι σημαντικό να τα αναφέρουμε εδώ, πιστεύω, σε αυτή την ομάδα. της Επιτροπής Απασχόλησης. Διότι ανησυχώ για κάτι. Ανησυχώ διότι πιστεύω ότι παρόλο που έγιναν ανεπίσημες διαπραγματεύσεις παρόλα αυτά έχουμε αυτή την εκκρεμότητα το πώς εκπροσωπείται η Επιτροπή Απασχόλησης Διαπραγματεύσεις αυτό το θέμα ίσως δεν το γνωρίζουν όλοι αυτό στη συνεδρίαση των συντονιστών που αντικαθιστούσα τη Γιούτα ετέθη το ζήτημα αυτό του Προέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης και της παρουσίας του Ο Τόμας Χέντελ δυστυχώς από ό,τι μάθαμε ε, έχει προβλήματα, το ευχόμαστε να καλυτερεύσει η κατάσταση. Δεν είχε προσκληθεί προσωπικά ο Τόμας Χέντελ ε, δεν έλαβε προσωπική πρόσκληση, προσεκλήθη ως πρόεδρος. Και όταν δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη την Επιτροπή μας μάλλον, πάντα έχουμε ε, έναν ε, προσωρινό αναπληρωτή πρόεδρο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής για να εκπροσωπούμεθα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε τώρα. διότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Κατά πόσο συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Δεύτερο ερωτηματικό. Το κείμενο, αυτό καθε αυτό. Οι ανεπίσημοι τριμερείς διάλογοι έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ψαχνόμαστε στο σκοτάδι. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Εδώ δεν είναι ξεκάθαρη η συνολική εικόνα και θα ήταν καλό πριν τη διάσκεψη των Προέδρων πριν δώσει η διάσκεψη των Προέδρων την άδεια στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπογράψει τη διακήρυξη στο Γκέτεμποργκ εμείς εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εξετάσουμε το κείμενο. Αυτό είναι το δεύτερο διαδικαστικό θέμα. Για το περιεχόμενο τώρα, από αυτά που είπατε, βλέπω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Διότι νομίζω ότι είναι σημαντικό να σημειώνεται πρόοδος στον κοινωνικό τομέα. Υπάρχουν προσδοκίες από το λαό. Και έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στο τριπλό α που ανέφερε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Ζιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση στην Ένωση. Συγχαρητήρια στους διαπραγματευτές. Συμφωνώ με τη Μάρια Ζωάου. Αν η διατύπωση στο πρώτο τμήμα της διακηρύξεως οδηγήσει σε κάποια ρεσιμότητα τότε ίσως διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο. Δηλαδή να υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες και να μην έχουμε ελάχιστα αποτελέσματα. Και εδώ είναι θέμα εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στα ευρωπαϊκά εγχειρήματα. Και αν συμβεί αυτό που προανέφερα, αυτό είναι το χειρότερο. Να υποσχόμεθα πράγματα χωρί να τηρούμε τι υποσχέσει, λόγω αιρεσιμότητα που αναφέρεται στο κείμενο, τότε επιδεινώνουμε την κατάσταση και δεν τη βελτιώνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Πυρίνσκι έχει το λόγο. Και βέβαια και όποιος άλλος θέλει μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να με βοηθήσετε σε κάτι. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Έφυγε ο κύριος Κάσα από τη συνεδρίαση. Και εγώ ήθελα να του απευθυνθώ, να πω κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που ανέφερε. Αν μπορείτε να διαβιβάσετε Α, Νάτος. Νάτος καλώς τον ε, κύριε Κάζα. Πήγα να φορτώσω με πρόσθετο καθήκον την πρόεδρο και ευτυχώς τη γλιτώσατε από αυτό. Επανέρχομαι σε αυτά που λέγατε, κύριε Κάζα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω σε αυτή τη φάση όπως είπατε κι εσείς. Εστιαστήκατε ουσιαστικά στο αν αξίζει τον κόπο να καταστρέψουμε ένα τέτοιο τεράστιο οικοδόμημα που δημιουργήθηκε με τέτοια προσπάθεια. Να το αντιστρέψω το ερώτημα. Γιατί το Συμβούλιο ξαφνικά αποφάσισε ότι πρέπει να βάλει αυτή τη λέξη μέσα. Δεν θα πρέπει να ζητήσουμε το Συμβούλιο να σκεφτεί τα επιχειρήματα που προβάλλατε εσείς. Αυτή είναι η λέξη κλειδί για το Συμβούλιο. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να μπούμε στην ουσία της επιχειρηματολογίας του Συμβουλίου. Γιατί, γιατί θέλω αυτή τη λέξη. Όπως είπε και η Μαρία Ζωάου, σοβαρή αιρεσιμότητα, δεύτερον, ποιοτική ε, αποδυνάμωση του πολιτικού μηνύματος. Και εγώ θα εισήγαγα και τρίτο επιχείρημα προβάλλοντας αντίρρηση στη λέξη would. Δεν είναι γεγονός από νομική σκοπιά. Δεν είναι νομική αναγκαιότης το ότι πολλές από αυτές τις 20 αρχές χρειάζονται κάποια νομοθετική εφαρμοστική πράξη. Δηλώνω τα γεγονότα αυτά τα κείμενα απαιτούν κάποιου είδους δράση. Το would θα γινόταν κάτι. Τι σημαίνει το would. Το would είναι, δεν έχει νόημα σε αυτό το πλαίσιο. Κύριε Κάζα, θα σας παρακαλούσα να αναγνωρίσετε ότι αυτή η εισαγωγή αυτής της λέξης, σε αυτή τη φάση μετά την σύνταξη κειμένου, το οποίο επεξεργάστηκαν επί μακρών συνάδελφοι, ξαφνικά. Να εμφανίζεται αυτή η λέξη και να ξεκινά ε, νέες διαπραγματεύσεις. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ανεύθυνο. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Κάσα. Έχει το λόγο, όπως προανέφερα, Θέλω να μιλήσουν και άλλοι και μάλιστα περισσότερο από μένα. Μου ετέθη το ερώτημα όμως. Δεν ξέρω αν γνωρίζει ο κύριος Πυρίνσκι ότι εμείς αποφασίσαμε προκαιρού, πολλού καιρού, ότι ή δυνατόν δεν θα αλλάξει λέξη τίποτα από το πακέτο, διότι θα καταρρεύσει το πακέτο ενδεχομένω. Αν το Συμβούλιο θέλει να, να προβάλλει αντιρρή σε πολλά άλλα σημεία, σε πολλά άλλα πράγματα, που, είναι πολύ σοβαρά για το Συμβούλιο, που δίνει την ευκαιρία με τη λέξη αυτή να το κάνει. Α είμαστε ειλικρινεί. Όλοι γνωρίζουμε, οι σέρπα γνωρίζουν. Είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα. Τι προσπαθώ να σας πω. Η λέξη would είναι τόσο σημαντική για μας, τόσο που ενδεχομένως να θέσει τέρμα στην όλη διαδικασία. Για μας του ΕΛΚ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν το επιτρέψω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι εκείνο που συνήθω θέτει τροχοπέδι και σταματάει του άλλου. Είμαι πολύ δημοκρατικό και συντονιστή, όπω ξέρουν και οι συνάδελφοι. Αλλά τώρα, σαν αφορά αυτή τη σημαντική στιγμή, τη μοναδική αυτή ευκαιρία που είναι sui generis, εγώ θα διαπραγματευόμουν με θετικό πνεύμα. Δεν θέλω να είμαι αρνητικό. Α είμαστε θετικοί. Ας προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ε, κατάσταση, να μην γίνει διαπραγμάτευση μονόδρομος, μην είμαστε μονόχνοτοι. Η κυρία Λάμπερτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ απηχώ αυτά που ακούστηκαν για τη συμμετοχή της Επιτροπής Απασχόλησης. Έπρεπε να σπρώξουμε για να μπούμε, ούτως υπήν και θέλω να διατηρήσουμε το χώρο μας εντός της διαδικασίας. Και είναι κάτι που θα επανέλθει στην Επιτροπή μας. Μετά τη διακήρυξη, τι θα κάνουμε με αυτό που θα δημιουργηθεί. Η διακήρυξη είναι κάτι υπέροχο, αλλά, αλλά, όπως είπαν και άλλοι, χρειάζεται και κάποια ουσία. Τώρα για τη διατύπωση τα επιχειρήματα μεταξύ του Σαλ και Μέι δίνανται και θα το πιο δεσμευτικό. Σε κάθε τριμερή διάλογο αυτά εμφανίζονται τα θέματα. Τώρα στη διακήρυξη χρειάζεται κάτι πιο θετικό η διατύπωση. Όταν τα κράτη-μέλη είναι σαφέστατα περί της αρμοδιότητας που έχουν σε αυτό. Κανένα κράτος μέλος δεν νομίζω δεν αναλαμβάνει κάποια δράση που θεωρεί ότι θα συμβάλλει στην κοινωνική Ευρώπη. Ίσως θεωρούν ότι είναι κάτι κοινωνικό για τη χώρα τους, αλλά αποτελεί κομμάτι του γενικού ευρωπαϊκού πλαισίου και τώρα θα πρέπει να εξετάσουν και τις διεθνείς υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι σαφέστατα συνδεδεμένοι στόχοι αυτοί με τον κοινωνικό πυλώνα. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η εξάλληψη της φτώχειας, ένας από τους βασικούς στόχους, και ταιριάζει βέβαια με τον κοινωνικό πυλώνα. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να είναι πιο ενθουσιώδη, πιο δυναμικά περί αυτών που πράττουν. Όπως είπα όμως, στον τριμερή διάλογο γνωρίζουμε ότι αυτό δεν διαπνέει πάντα αυτό, αυτό το στοιχείο του διαλόγου. Τώρα, την μετά διακήρυξη εποχή. Πρέπει να σκεφτούμε και το πώς το Κοινοβούλιο θα παραμείνει εντός της διαδικασίας. Ίσως ελπίζουμε για κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά υπάρχει και η διάσταση της ήπιας πολιτικής που θα πρέπει να προωθούμε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπου η διακήρυξη φαίνεται κάτι πολύ πιθανό. Θα προχωρήσουμε κάποια θεσμικά όργανα, ελπίζω και τα τρία θεσμικά όργανα να εκπροσωπούνται και να έχουν πολυπληθεί αντιπροσωπεία. Το Ευρωκοινοβούλιο βέβαια είναι το άμεσα ερετό ευρωπαϊκό ε, κομμάτι. Σε αυτή την Επιτροπή και εντός του Κοινοβουλίου πρέπει να δούμε πώς θα παίξουμε τον ρόλο που μας αρμόζει. Να μην παραμείνει άσκηση σε πιχάρτου η διακήρυξη. Δεν ξέρουμε αν το θα το έχουμε πάνω σε περγαμηνή με καλλιγραφία ή θα βρούμε κάποια άλλη εναλλακτική χρειάζεται να είναι κάτι παραπάνω από τη γραπτή διακήρυξη. Θα πρέπει σε, σε επίπεδο επιτροπής ή σε επίπεδο συντονιστών να το συζητήσουμε αυτό. Ευχαριστώ και κύριο Σούστερ. Μου φαίνεται πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Ο συμβασμός όμως θα πρέπει να έχει κάποια ουσία, κάποιο ουσιαστικό περιεχόμενο. Αλλιώς δεν είναι παραδεκτός ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να γίνουμε το φίλο οικής που τελικά να κρύψει το γεγονός ότι ορισμένοι δεν ε, μιλούν σοβαρά όταν μιλούν για κοινωνικό πυλώνα. Όταν διαγράφεται μια λέξη, συνήθως αυτή η λέξη έχει μεγάλη σημασία. Αλλιώς δεν υπάρχει και λόγος να διαπληκτίζεται κανείς τόσο καιρό για την ε, λέξη αυτή. Και καθώς διαβάζω το κείμενο, θεωρώ ότι αν θέλουμε οι αρχές αυτές να είναι αναγκαστικές, να είναι εκτελεστές, θα πρέπει να υπάρχει αναγκαία νομοθεσία. Αν όμως λέει θα πρέπει ή θα έπρεπε να ψηφιστεί έτσι και αλλιώς και τα λοιπά, τότε ανοίγουμε ένα μεγάλο παράθυρο για να μπορούν να φύγουν μερικοί. Θα πρέπει να πει το Συμβούλιο ότι εμείς εμένουμε στις αρχές και η εφαρμογή τους απαιτεί να ψηφιστούν στο κατάλληλο επίπεδο. Αυτό θα ήταν το σωστό. Αν μπει αυτό το good αμέσως ξυπνά την υποψία ότι κάποιες χώρες δεν μιλούν σοβαρά όταν τα λένε αυτά τα πράγματα. Ότι θα το κάναμε, αλλά τελικώς δεν θα το κάνουμε. Και πολύ σωστά είπε η Μαρία Ζωάου ότι είναι ένα σημαντικό θέμα αξιοπιστίας ευρωπαϊκής αξιοπιστίας. Δεν βλέπουν καθαρά ότι υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές απαιτήσεις που πρέπει να ρυθμιστούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε διακήρυξη δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αποδυνάμωση του μηνύματος, τουλάχιστον εκεί θα πρέπει να μπει ένα ξεκάθαρο κείμενο όπου δεν έχει καμία θέση βεβαίως αυτός ο υποθετικός λόγος. Ευχαριστώ, Κλοντ Ρολάν. Ευχαριστώ. Πράγματι. Μας απασχολεί το θέμα και έχει ρόλο να παίξει η Επιτροπή Απασχολήσεως. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι να υπάρξει η διακήρυξη αυτή. Προφανώς έχει δύο στοιχεία αφενός να είναι χρήσιμη, αποτελεσματική επομένως σε συγκεκριμένα πράγματα. Έχει όμως και έναν έντονο συμβολισμό και γνωρίζουμε ότι στην πολιτική ο συμβολισμός έχει σημασία. Ο συμβολισμός βαραίνει στα πράγματα, έχει, έχει ένα ρόλο, έχει ένα βάρος. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να απογοητεύσουμε τον κόσμο. Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Πρώτο, η έλλειψη σαφήνειας. Όμως ακόμα περισσότερο, αν τελικώς αποδειχθεί αποτυχία και δεν υπάρξει διακήρυξη, εγώ νομίζω ότι τότε η απογοήτευση θα είναι τεράστια των ανθρώπων αυτών που αναμένουν κάποια βήματα πρόοδου της κοινωνικής Ευρώπης. Εγώ θα προτιμούσα το Συμβούλιο να μην έχει την θέση αυτή που έχει. Αλλά είναι γεγονός ότι την έχει. Δυστυχώς θα έλεγα. Αλλά έτσι είναι και οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη. Δεν χρειάζεται να σα εξηγήσω εγώ στου παρόντες που γνωρίζετε πολύ καλά τα στοιχεία αυτά. Μια διαπραγμάτευση πάνω σε μια διαφορά τι σημαίνει. Υπάρχει το ένα μέρο που έχει μια θέση α, άλλο μέρο το οποίο έχει μια θέση β και εν τέλει για να λειτουργήσει χρειάζεται μια λύση γ. Ούτε α, ούτε β, αλλά γ. Και νομίζω ότι εν προκειμένου έχουμε μια θετική αρμοδιότητα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ, κυρία Μέλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι για την συνάντηση αυτή που γίνεται γύρω από την σημειολογία του κειμένου. Καιρό είχα να συμμετάσχω σε τέτοια σημειολογική συνάντηση που μας κάνει να ξεχάσουμε και την ουσία του θέματος και της ε, διακήρυξης. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη δυσκολία για τον ίδιο τον πυλώνα και για τις 20 αυτές αρχές. Είναι αρκετά ε, σημαντικό. Πρόκειται για μια φυσιολογική διακήρυξη προγραμματικού χαρακτήρα θα έλεγα εγώ, οποιοδήποτε υποψηφίου σε οποιαδήποτε χώρα. Πολύ ευρεία θα δώσει πλεονεκτήματα σε όλους, όλα τα πράγματα θα γίνουν καλά. Βεβαίως τα τρία τέταρτα των υποσχέσεων δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, διότι δεν είναι δυνατόν και ιδίως στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όποια και αν είναι τελικώς η διατύπωση του προημίου, το προήμιο αυτό εμπεριέχει και παράδοξα. Και η κυρία Λαμπέρ ανησυχεί για την συνέχεια που θα δοθεί στην διακήρυξη. Εγώ νομίζω ότι η διακήρυξη ήδη εμπεριέχει την προγραμματισμένη της αποτυχία, διότι λέει ότι θα γίνουν ε, σεβαστές οι αρχές, ότι η ζώνη ευρώ θα ε, είναι κυρίως αυτή που, που στοχεύεται αν και έχει μεγαλύτερη ενέργεια από τη ζώνη μη ευρώ θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κρίση ενώ θα έπρεπε ίσως να δοθεί άλλη απάντηση με την έννοια ότι διαφορετικές ευρωπαϊκές δομές ευθύνονται εν μέρη για το γεγονός ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να μην έρχεται. Γνωρίζετε ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Γνωρίζετε, τα είπαμε αυτά και στην Κροατία, για το dumping θα αρκούσε να καταργηθεί η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και για να υπάρξει μια ευθυγράμμιση των κοινωνικών συστημάτων για να εξαφανιστεί το dumping ενώ η διαφορά των βασικών μισθών είναι μέχρι και δεκαπλάσια. Αυτά είναι στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προήμιο και που τελικώς Εν τέλει, οι Ευρωπαίοι πέραν από τους συμβολισμούς αναμένουν αυτά αποτελέσματα. Να υπάρξει απασχόληση. Να μην υπάρχουν αναλογίες της τάξης του 25% του εργατικού δυναμικού να είναι στην ανεργία με βαρύτατες επιπτώσεις στα κοινωνικά συστήματα διότι οι άνθρωποι που δεν εργάζονται ούτε αμείβονται ούτε εισφέρουν κοινωνικά, άρα είναι καταστροφική η εξέλιξη και για τις συντάξεις και για την κοινωνική πρόνοια. Προτείνω λοιπόν να θεωρήσετε ότι ώρες είναι οι μεγαλόστομες διακηρύξεις, αλλά θα έπρεπε να ασχοληθεί κανείς περισσότερο με την ουσία. Ευχαριστώ. Κύριε Κάσα, θέλετε και πάλι το λόγο επιθυμώ να σας υπενθυμίσω ότι δεν συναντώμεθα εδώ για να αλλάξουμε τίποτα. Πρόκειται για παρουσίαση του κειμένου. Όπως ίσως έχετε ακούσει, υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι αντιτίθεται καν στην έγκριση της διακήρυξης. Χρειάζεται λοιπόν λίγη προσοχή. Υπάρχουν πράγματα που δεν μου αρέσουν ως λαϊκό κόμμα. Αλλά είμαι διατεθειμένος να κάνω μια παραχώρηση δεν είναι εύκολο και η Επιτροπή, το γνωρίζετε όλοι, δεν θα έχει τη δυνατότητα η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή να αλλάξει την διατύπωση. Αυτό έλεγα και από την αρχή. Κάναμε έκθεση, συζητήσαμε τα πράγματα αυτά. Δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την ουσία. Διότι αυτή τη στιγμή αρχίσουμε να συζητούμε την ουσία και το τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ουσία, ανοίγεται την πηξίδα της Παρδόρας όλοι θα αρχίσουν να θέλουν να αλλάζουν κάτι, μια παράγραφο, ε, μια φράση. Μπλέξαμε τότε. Προσοχή λοιπόν, η διαδικασία δεν ήταν η καλύτερη, συμφωνεί, η καλύτερη που μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Κοινοβούλιο. Ζητήσαμε και από την Προεδρία, ζητήσαμε και από έναν εκπρόσωπο κάθε πολιτική ομάδα. Αν τελικώ δεν εγκριθεί, λοιπόν πολύ. Αυτό έχουμε τώρα όμω μπροστά μα. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να το κλείσουμε. Άρα, προσοχή και ας μην περιπλέξουμε τα πράγματα περισσότερο από όσο είναι ήδη περίπλοκα. Να με συμπαθάτε που πήρα το λόγο και για τρίτη φορά, αλλά έπρεπε να τα πω τα πράγματα αυτά. Άλλος επιθυμεί να δευτερολογήσει ο κύριος Πυρίνσκι. Η πρώτη μου ε, παρέμβαση ήταν ερώτηση και όχι τοποθέτηση. Η κυρία Λάμπερτς είπε ότι περιοδικά επανέρχεται αυτή η δυσκολία με το Συμβούλιο, με τις διατυπώσεις του Σαλ και του ΜΕΙ, οριστικής ή υποθετικής δηλαδή. Αλλά προκειμένου δεν πρόκειται για Σαλ και ΜΕΙ, διότι το κείμενο για αυτούς είναι καθαρό. Οι αρχές και τα δικαιώματα για να είναι νομικός εξαναγκαστά χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα ή νομοθεσία που θα εγκριθεί στο κατάλληλο επίπεδο το Συμβούλιο βάζει μέσα τη λέξη would require, που θα απαιτούσε την νομοθέτηση στο κατάλληλο επίπεδο. Η ουσία εδώ, εν προκειμένου, είναι να δείξουν πολιτική βούληση. Και για να δείξουν πολιτική βούληση, εν προκειμένου, για ότι 20 αυτές αρχές, εν ευθέτω χρόνο και σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις επιθυμίες των κυβερνήσεων και κοινοβουλίων θα βρεθεί, θα μπορέσει να νομοθετηθεί. Ο κ. Ρολά είπε ποια θα είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση. Να βγει η διακήρυξη με αυτό το good require ή να μην βγει καθόλου. Εγώ νομίζω ότι μια ιονή διακήρυξη που εκφράζει μια προσμονή αλλά αδύνατη πολιτική βούληση είναι και χειρότερο από το να μην υπάρξει διακήρυξη. Και να είναι καθαρό ποιος τάσεται υπέρ τίνος. I think some... νομίζω πως κάποιον ξέχασα που ζήτησε το λόγο. Okay, uh, I have not. Uh, Όχι. Ωραία. Τότε Μήπως υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Επιτροπή. Σα Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω δύο λόγια. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ του ΣΕΡΠΑ για την εργασία τους που είναι εξαιρετική και που μας φέρνει πολύ κοντά σε συμφωνία για το κείμενο που είναι πολύ καλό. Είπαν οι ΣΕΡΠΑ, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω, ότι το γεγονός ότι οι αρχές είναι τώρα επιτάπητος και ότι έχουν συμφωνηθεί από τα κάτι μέλη ακόμα και από αυτά που ήταν πολύ αρνητικά για την ιδέα με, ακόμη της κοινωνικής σύγκλησης είναι κάτι που το, είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι νομίζω περίπλοκο ε, και βεβαίως αν ε, μου επιτρέπετε να κάνω κάποιες επεξηγήσεις αυτό το εκτιμώντας είναι ένα εκτιμώντας που μιλάει για τα εφιστάμενα δικαιώματα. Και δεν αμφισβητεί κανείς στο Συμβούλιο το γεγονός ότι αυτά τα εφιστάμενα δικαιώματα είναι νορμικά εφαρμοστέα. Άρα η συζήτηση αφορά τις νέες αρχές, τις αρχές για τις οποίες σήμερα δεν υπάρχει νομική εφαρμογή επειδή δεν υπάρχει ε, οδηγία, επειδή τα κρατημέλη δεν έχουν εθνική νομοθεσία. Υπάρχουν κάποιες αρχές όντως που είναι νέες. Νέες με την έννοια ότι σήμερα δεν υπάρχει νομική εφαρμογή. Αυτό που θέλουν να κάνουν τα κρατημέλη, νομίζω, ε, με βάση τα όσα είπαν στην Κορεπέρ, ήθελα να καταστήσουν σαφές ότι αυτά που περιλαμβάνονται στις αρχές δεν θα δημιουργήσουν αυτά καθε αυτά νομικά δικαιώματα. Δεν είναι δηλαδή αυτόματο. Χρειάζεται νομοθεσία είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο, ώστε αυτά τα δικαιώματα να είναι εφαρμοστέα. να είναι εξαναγκαστά. Ε, αυτή είναι η έννοια που θέλουμε να επιμείνουμε και έτσι κάποια κράτη-μέλη πρόσθεσαν την, το good πρότειναν να προσθεθεί το Wood. Δεν είναι καλή διατύπωση, συμφωνώ. Δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι προαιρετικό αλλά αν ε, τελικά διαβάσει κανείς τη φράση, ε, αντιστοιχεί στο μήνυμα που θέλαμε να διαβιβάσουμε, ότι δηλαδή αυτές οι νέες αρχές όπου δεν υπάρχει ακόμα εθνική νομοθεσία ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, χρειάζεται να ληφθούν κάποια μέτρα είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ένωση, ενωσιακό. Αυτή είναι μια σύντομη εξήγηση της συζήτησης και εγώ είμαι ο πρώτος που συμφωνώ πως η διατύπωση που επελέγει από τα κάθε μέλη δεν είναι κομψή και ότι ε, θα πρέπει να προτείνουμε νέα και διαφορετική χάρη σε κοινέ προσπάθειες με τους ΣΕΡΠΑ να μετατρέψουμε το wood σε Sud. και έτσι να μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Περισσότερο είναι προσωπική μου παρατήρηση, γιατί αν δείτε τις άλλες παρατηρήσεις, ε, παράγραφους μάλλον στο κείμενο, κάποιες φορές δεν είναι καλά διατυπωμένα. Οπότε μπορεί να πει κανείς γιατί επιμένεις πάλι σε αυτή την συγκεκριμένη επιλογή ε, λέξεων. Ε, το θέμα είναι αν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, μήπως διατρέχουμε το κίνδυνο να το διαλύσουμε όλο γιατί ήταν μεγάλη η πρόκληση και μεγάλη επιτυχία που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και βρήκαμε σχεδόν συμφωνία και ότι συζητάμε μόνο για μία λέξη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε. Υπάρχει κίνδυνος να διαλυθεί όλη η συμφωνία και να ξαναρχίσει η συζήτηση για τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ελπίζω λοιπόν πως αυτή μου η εξήγηση θα χρησιμεύσει για τις δικές σας ε, διαβουλεύσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ας επανέλθουμε στο ΣΕΡΠΑ τώρα να αρχίσουμε τον κύριο Φαντεκέντελερ. Ποια είναι τα δικά σας σχόλια από την σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας τις απόψεις για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Όπως είπα στην αρχή, πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατάσταση και το ότι ήρθαμε να σας ενημερώσουμε στη μέση μια διαδικασία τριμερού διαλόγου είναι πάλι περίεργο, αλλά είναι νομίζω γέννη καλή πρακτική και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε να το επαναλάβουμε και σε, άλλες, σε, σε άλλους φακέλους, σε άλλα θέματα. Η, το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ έχει τις δικές του θέσεις και τη δική του δυναμική ε, που διαφέρουν από αυτές του Κοινοβουλίου και αυτό είναι σαφές για όλους μας νομίζω πλέον. Κατά κάποιο τρόπο πλησιάζουμε στο τέλος και δεν θα πρέπει να χάσουμε την επερχόμενη ευκαιρία. Οπότε θα χρειαστεί να βρούμε, όπως είπε σωστά και ο κ. πολύ ρεαλιστικά, ότι θα πρέπει να βρούμε δηλαδή κάποια λύση. Όχι ότι αφήσουμε το κείμενο κενό νοήματος. Όχι, αυτό το προσέχουμε πολύ. Όταν ε, πρόκειται για το θέμα των ΣΕΡΠΑ ως τρίτος ΣΕΡΠΑ, Εγώ προσωπικά θα ήθελα η, η, πρόσκληση να μην είναι ad αλλά ad Και επίσης ε, το κείμενο της συμφωνίας θα πρέπει να ξανάρθει στην Επιτροπή πριν ληφθεί απόφαση. Όσον αφορά την διάσκεψη κορυφής, είμαι τη άποψης, όπως και η κυρία Ροντρίκη, ότι πρέπει να έχουμε μια ισχυρή εκπροσώπηση στη διάσκεψη κορυφής ε, και επιθυμούμε ε, να στρίξουμε λοιπόν, να, ε, να υποστηρίξουμε αυτό το έγγραφο. Τώρα αφορά το συμβολισμό του γράφου αυτού, βεβαίω το βαθμό του συμβολισμού είναι σημαντικός. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το συμβολικό, τη συμβολική μάλλον μορφή πτυχή του, της διακήρυξης. Χαίρομαι που το Ευρωκοινοβούλιο είναι στο διαπραγματευτικό τραπέζι για αυτό το θέμα, αλλά όπως είπε και σωστά η κυρία Λάμπερτς, έχουμε ένα έργο και ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση να προβληματιστούμε για το ρόλο μας όταν ε, πρόκειται για την μετά ε, ε, φάση, δηλαδή τη φάση μετά την προκήρυξη. Έχουμε και εμείς μέλλον για την υλοποίηση ε, του κοινωνικού πυλώνα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σχετική συζήτηση και μάλιστα σύντομα. Κύριε Ροντρίγκε, συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι ε, Όσον αφορά τον τρόπο ανάμεξης τη Επιτροπή ΕΜΠΛΟ, θα ήταν καλύτερο ο πρόεδρο ή ένα αντιπρόεδρο να αντιπροσωπεύσουν το σύνολο τη Επιτροπή. Ωστόσο, όπω μπορείτε να δείτε, φτάνουμε στο τέλος και γι' αυτό το να παραμείνει η Επιτροπή Απασχόλησης μέσα στην διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η συζήτηση ήταν πολύ βοηθητική και ε, εάν καταφέρουμε να γίνει αυτή η διακήρυξη στην, στην διάσκεψη κορυφής του Γκέτεμπορ, το Κοινοβούλιο θα στηρίξει με όλες του τις ομάδες την διακήρυξη αυτή και γιατί αυτή στέλνει πολύ σημαντικό μήνυμα. Να υπογραμμίσω ότι θα μπορούσαμε σε αυτό το τριμερί να καταφέρουμε να πετύχουμε τη σημαντική αναγνώριση των δικών μας θέσεων, ειδικά όσον αφορά το ρόλο των κοινωνικών εταίρων που αναγνωρίστηκε πλήρως και δεύτερον όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής αυτού του πυλώνα που θα πρέπει να αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Πολύ σημαντικές διευκρινήσεις αυτές. Να τελειώσω με το τελευταίο εκκρεμές θέμα. Ε, Όντω, ε, όπω υπεγραμμίζουν κάποια μέλη της Επιτροπής, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο μια θέση, μια εργασία. Είναι η πρόθεση, η στάση που διέπουν την διακήρυξη που ποτίστε θα γίνει στο Γκέτεμπορκ. Και δεν μπορούμε να δώσουμε την εντύπωση ότι με αυτή τη ε, διακήρυξη Ανακοινώνουμε 20 καλές αρχές για να βελτιωθούν ε, οι συνθήκες εργασίας ε, των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά ταυτόχρονα λέμε στην ίδια διακήρυξη ότι μας αρέσουν αυτές οι αρχές, αλλά ε, πρέπει ακόμα να συζητήσουμε αν θα πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Δεν μπορούμε να στέλνουμε τέτοιο μήνυμα. Πιστεύω λοιπόν πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πει ότι αυτή η λέξη would δεν μπορεί να σταθεί εδώ. Δεν γίνεται να το δεχτούμε για αυτό το λόγο. Όμως όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση και αυτό συμβαίνει συχνά στους τριμερείς, ο ρόλος της Προεδρίας είναι να βρει μια καλή συμβαστική. Και σε αυτό είμαστε ανοιχτοί. Αλλά εξηγήσαμε σαφώς και νομίζω πως ε, πρόκειται για απλή πολιτική λογική να μην διακηρύσεις κάτι και μέσα στο ίδιο κείμενο να ανακοινώνει ότι ακόμα είναι υποσυζήτηση το αν θα εφαρμοστεί ή όχι. Γιατί έτσι δημιουργείς εντυπωσει. Mr. Κάσα. Ε, κύριος Κάσα. Ε, κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ μετά όσα είπε η κυρία Ροντρίκη. Δεν αντιπροσωπεύει το Κοινοβούλιο μαζί με τον Τόμα, αντιπροσωπεύει μέχρι στιγμή την ομάδα μας. Ε, η δική της θέση δεν είναι η θέση της πλειοψηφίας. Προσέξτε λοιπόν όταν κάνουμε δηλώσεις. Δεν έχει να κάνει με την προσωπική δόξα οποιοδήποτε εδώ. Θέλουμε να είναι μια προσπάθεια που θα μας ενώσει και που θα να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν να είναι από την ίδια πλευρά. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να αρχίσουμε πάλι να τα συζητάμε. Δεν είναι δεσμευτική αυτή η δήλωση, οπότε ας μην υπερβάλλουμε. Όταν λοιπόν πρέπει να διαπραγματευτούμε ε, για αυτά τα οποία είπε η κυρία Ροντρίγκε, να πούμε ότι αντιπροσωπεύεται, να θυμίσουμε ότι αντιπροσωπεύεται ολόκληρη την Επιτροπή και όχι μόνο κάποιου. Η κυρία Ιονγκέριου. Διερωτώ με. Μήπως ο κύριος Κάζα εννοεί τελικά ότι πρέπει να ψηφίσουμε για το αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί όχι, γιατί αν λέτε ότι η κυρία Ροντρίκης δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία της Επιτροπής, Δεν ξέρω πώς ε, το μετρήσατε ή αν ε, θα πρέπει να έχουμε ψηφοφορία να κάνουμε γι' αυτό. Για μένα είναι σημαντικό και νομίζω πως αυτό είναι και ο λόγος ύπαρξης όλης αυτής της ε, προσπάθειας, ότι δηλαδή όχι μόνο να είναι καλή η συνεδρίαση στο Γκέτεμπορκ, αλλά να έχουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό συμβολικό μήνυμα ε, που θα στείλουμε στους πολίτες της Ευρώπης. Εκείνη τη μέρα στο Γκέτεμπορκ και από εκεί και στο εξή. Αν θέλετε να ψηφίσουμε ωστόσο, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα. Ναι, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε όχι. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε γιατί αν ψηφίσουμε, όχι, δεν θα έχουμε την, ε, την, ε, την ε, δήλωση, την, την προκήρυξη. και οι Σέρβας το ξέρουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ψηφοφορία γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Θα ήταν κακό, αρνητικό για όλους και για τους σοσιαλιστές γιατί θα έχετε και το Προεδρείο για να το δείξετε ακόμη πιο σπουδαίο και να γίνει πιο σημαντικό. Εγώ δεν το είπα εγώ ο ίδιος. Η κυρία Ροντρίγκες ανέφερε αυτό το πρόβλημα του Γουντ. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι προσπαθήστε να μεταφέρετε την πλειοψηφία αυτής τη επιτροπή και του Κοινοβουλίου και όχι μόνο την ε, προσωπική σας γνώμη. Γιατί όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί λοιπόν, όμως να παραμείνει προσωπική άποψη πρέπει να αντιπροσωπεύει το Κοινοβούλιο. Αυτό θα επιθυμούσα. Δεν θέλω ψηφοφορία, δεν θέλω να ανοίξουμε τίποτα γι' αυτό, γιατί έχουμε συμφωνία τώρα. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γίνει αυτή η συζήτηση και να ε, βοηθήσουμε μόνο τους λαϊκιστές που θα χαρούν με, τη... με αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Έτσι κι αλλιώς με τόσους λίγους εδώ δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Θέλετε το λόγο, κύριε Πυρίνσκι, όχι. Εγώ νομίζω πως είναι φανταστικό που έχουμε συζήτηση για αυτό το θέμα. Το κοινωνικό πυλώνα και την κοινωνική ατζέντα. Και μάλιστα όταν πλησιάζουμε τις, ευρωπαϊκές, τις ευρωεκλογές. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ατζέντα όλοι, είτε είναι οι σοσιαλιστές, είτε είναι το ΕΛΚ, είτε είναι οι φιλελεύθεροι, μια ατζέντα με κοινωνικό περιεχόμενο. Ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με τεχνικά θέματα που οι ψηφοφόροι και οι πολίτες ε, δεν βρίσκουν ενδιαφέροντα. Αυτό εδώ το θέμα αφορά τη ζωή τους, την ε, αξιοπρέπειά τους, αφορά την δικαιοσύνη και αυτό είναι πραγματικά ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα ήθελα λοιπόν να επιτεθούμε εναντίον του επειδή δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση αυτή τη στιγμή για την ακριβή διατύπωση. Είμαι βεβαία πως η συζήτηση θα συνεχιστεί ατύπως. Αλλά ίσως να χρειαστεί να επανέλθουμε και τύπης με κάποιο τρόπο, αλλά πάντως να μην αφήσουμε αυτό να μας φάει την ενέργεια που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της συνεδρίασης, γιατί είμαστε ενωμένοι σε τόσα θέματα και αυτό είναι σημαντικό και αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα επανέλθουμε στο θέμα της ε, διατύπωσης, μπορεί να το κάνουμε. Αλλά ας μην αφήσουμε αυτό το σημείο να μας παραλύσει. Θα έχουμε πολύ ισχυρή εκπροσώπηση στο Γκέτεμποργκ, θα έχουμε ισχυρή εκπροσώπηση που δείχνει ότι είμαστε ενωμένοι και μόνο το γεγονός ότι έχουμε συζήτηση, πρόταση, διαδικασία και κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης. Δεν μπορώ να τελειώσω αυτή τη συζήτηση με μεγαλύτερη ακρίβεια ακόμη, γιατί είδαμε πως υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ε, δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο βαθιές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε Και τούτο λεχθέντος να πω επίσης του ΣΕΡΠΑ που ίσως να χρειαστεί να ξανασυνεδριάσουμε. Ελπίζω πως θα πείτε ναι στην πρόσκληση αν θελήσουμε να ξανασυνεδριάσουμε. Ας προχωρήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή η συνεδρία συνεδρίαση στο Γκέτεμπορκ να σημαίνει κάτι. Και από την πλευρά της Επιτροπής, να βεβαίως ποτέ δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί είμαστε η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για αυτή την ε, ε, τα θέματα και, δεν θα ησυχάσουμε αν δεν αντικρουσοποιηθούμε στο Γκέτεμπορκ. Και βεβαίως οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να το αφροντίσουν αυτό. Ίσως να είναι μια, ένας αγώνας σε μια μάχη που θα δώσουμε και θα χάσουμε. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να την κάνουμε αυτή τη ε, μάχη. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και θα αλληλοενημερωνόμαστε. Ίσως λοιπόν να γίνουν και περισσότερες συνεδριάσεις και να πρέπει να τις προγραμματίσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε <clears throat> και για την σημαντική σας υποστήριξη και για τα δηλώσεις σας. Η σημερινή μας συνεδρίαση λοιπόν ε, ολοκληρώθηκε.